κάνει ταχύτατα προτάσεις έτσι ώστε τα προγράμματα Εράσμος και Λεωνάρντο να λειτουργήσουν το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ κύριε Πεγιόν. Ας περάσουμε τώρα στη δεύτερη ανακοίνωση του Προεδρείου. Πρόκειται για μια διόρθωση. Σας ανακοινώνω ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς μετέφερε τις εξής τροποποιήσεις σε δύο κείμενα τα οποία ενεκρίθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις προϋποθέσεις για την με τις ρυθμίσεις ασφαλείας για τα αυτοκίνητα οχήματα και τα α, σειρώμενα από αυτά. Επί τη βάση του 216 παράγραφος 4 τέτοιου είδους διορθώσεις θεωρούνται δεκτές εκτός και αν μέσα σε 48 ώρες μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 βουλευτές εκφράσουν την αντίθεσή τους. Οι διορθώσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Είκοσι δευτερόλεπτα μόνο. Κάθε μήνα είμαστε υποχρεωμένοι ευτυχώς να ερχόμαστε εδώ στο Στρασβούργο και το κάνουμε με ευχαρίστηση. Θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση όμως στην Προεδρία έτσι ώστε να μας μεταφέρει την άποψή μας αυτή και προς την Επιτροπή. Θα πρέπει νομίζω σε επίπεδο δυνατοτήτων μετακίνησης να απλοποιηθούν τα πράγματα. Εμείς η Ιταλική Αντιπροσωπεία και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, δεν καταφέρνουμε να έχουμε απευθείας πτήσεις είτε από τη Ρώμη είτε από άλλες πόλεις προς το Στρασβούργο. Είμαστε υποχρεωμένοι να ταξιδεύουμε για μια ολόκληρη μέρα. Χτες ταξίδευα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νομίζω ότι πρέπει να πάρετε κάποια μέτρα, να απευθύνετε το αίτημά μας προς την ΕΦΡΑΝΣ, προς το γαλλικό κράτος, σε βάση περιπτώσει να υπάρξουν κάποιες προτάσεις για να μπορούμε να φτάνουμε στην πόλη του Στρασβούργου χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία. Ευχαριστώ κύριε Αντινορό. Προφανώς και δέχομαι το ξεκάθαρο μήνυμά σας και η Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί να κάνει μεταφέροντας αυτή την ενόχληση που εκφράσατε σχετικά με την επιμελητία που δεν αφορά μόνο την Ιταλική αντιπροσωπεία. Βέβαια δεν θα γίνει συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό τώρα. Ε, περνάμε στις ψηφοφορίες. Αλφάνο. Μία παρατήρηση, Πρόεδρε σχετικά με αυτήν την ψευδοεκένωση που κάναμε στο Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Έγινε κάτι εκτός κανονισμού. Κανένας δεν μας ειδοποίησε στα γραφεία ότι έπρεπε να εκενώσουμε το κτίριο και εκτός Κοινοβουλίου ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε, δεν ήξερε τι να κάνει. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι λεφτά ξοδεύουμε σαν Κοινοβούλιο κάθε χρόνο για την ασφάλεια του Κοινοβουλίου και για τους κανόνες εκένωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι κανόνες λίγο πιο αυστηροί. Ευχαριστώ κύριε Αλφάνο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προέβλεψαν να ειδοποιηθούν όσοι ήταν εκεί μέσα στο κτίριο και οι βουλευτές μέσω των ε, υπεύθυνων ασφαλείας. Ήταν το μοναδικό που μπορούσαν να κάνουν. Εν πάση περιπτώσει τώρα περνάμε στις ψηφοφορίες, δεν ανοίγουμε άλλες συζητήσεις. Για την κυρία Κοπά τώρα, έκθεση της κυρίας Κοπά. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, δεκτή. Έκθεση Τίκαου, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Έκθεση Γκάλαχερ, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Avete votato tutti? Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Γίνεται δεκτή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Έκθεση Ρόιλ. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή έκθεση Ρόιλ. Έκθεση Οκονή. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Κυρία Ματίας. Έκθεση Ματίας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συγχαρητήρια κυρία Ματίας. Καβαντά. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή συγχαρητήρια στον κύριο Καβαντά το Ιρερ είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή συγχαρητήρια στον κύριο Τόιρερ Γκαρντίνη είναι υπέρ κατά αποχές συγχαρητήρια στον κύριο Γκαρντίνη ο Κονή επίσης ποιοι είναι υπέρ α συγγνώμη για μια στιγμή α Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό το πρώτο τμήμα. Θέτω σε ψηφοφορία τώρα. Το σύνολο της πρότασης τροποποιημένη. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος. Μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Κονή. Η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση Lightfried. Έχει ζητήσει το λόγο κύριο Lightfried. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να μιλήσω και θα επισημάνω κάτι. Νομίζω Μέχρι τώρα πάντα ταχτήκαμε ε, με το μέρος των ε, δημοκρατών. Όχι στην πλευρά των δικτατόρων και εκείνων που υπερασπίζονται, που πιέζουν μάλλον και αγνοούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι πολύ κρίσιμο. Πρόκειται για μια έκθεση με οικονομικά συμφέροντα και υπάρχουν κάποιες ε, αμφιβολίες το τι θα πρέπει να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ε, software ε, παρακολούθησης ε, δεν θέλουμε να το δώσουμε σε δικτάτορες γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να ελέγχουν το Twitter, το Facebook αυτά είναι ευρωπαϊκά προϊόντα τα οποία ε, μέχρι τώρα εστάλησαν μόνο μέχρι τη Βόρειο Αφρική. Στο μέλλον τα πράγματα θα αλλάξουν. Και το μόνο πρόβλημα σε όλο αυτό το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ελέγχουμε μετά την παράδοση των προϊόντων. Ίσως ε, με την επόμενη εκθεσή μας να μπορέσουμε να κάνουμε τον έλεγχο πριν από την παράδοση αυτών των προϊόντων. Αυτή είναι η παράκλησή μου αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστούμε συνάδελφε για αυτές τις εξηγήσεις σας. Πάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία η 52 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται πρόταση της ε, ως τροποποιήθηκε υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ε, εγκρίνεται ονομαστική κλίση ψηφίζουμε παρακαλώ έκλεισε ψηφοφορία. ευρύτατη η πλειοψηφία και για αυτή την έκθεση συγχαρητήρια λοιπόν έκθεση Φιντάντσα Ψηφίζουμε παρακαλώ υπέρ κατά αποχές ε, συγχαρητήρια στον κύριο Φιντάντσα εγκρίθηκε η έκθεσή του. Έκθεση Κοχ. Παράγραφος 4. Υπέρ παρακαλώ. Με ονομαστική κλίση. Συγγνώμη, το ξέχασα. Με ονομαστική κλίση. Ζήτησε να μιλήσει ο εισηγητής.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 με ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παράγραφος 26. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 μισό λεπτό. Για την 50 παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίθηκε με ευρύτατη ψηφοφορία 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Για την 54 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίθηκε και αυτή 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροποποιημένη πρόταση υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Έκθεση ΔΕΒΑ. Ε, μισό λεπτό. Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Παράγραφος 23. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Για το τρίτο τμήμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η παράγραφος 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 29. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και εγκρίθηκε. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Μα είναι η ίδια η πλειοψηφία όπως πριν. Αν θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο, ευχαριστώ να τον κάνουμε. Όχι, δεν θέλετε. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές γκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ψηφίζουμε ηλεκτρονικά δεύτερο τμήμα του 45 έκλεισε η ψηφορία και απορρίπτεται Δι ε, υπέρ παρακαλώ κατά Ψηφίζουμε για την αιτιολογική σκέψη D. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Ε, η πρόταση ψηφίσματος, το σύνολό της, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές ε, η πρόταση εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Ντέβα. Πάμε στην επόμενη έκθεση. Τσίμα. Τσίμα. Λοιπόν, Παράγραφος 36, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και απορρίφθηκε. Παράγραφος 39. Σε χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 40 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπέρ για το δεύτερο τμήμα κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 44 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 53 πρωτοτμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές ε, κατά ήτανε, ελέγχουμε για το δεύτερο τμήμα της 53, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίθηκε. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 70 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 70 ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίθηκε η 70. 73 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έκλεισε η ψηφοφορία και εγκρίθηκε. 74 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, αιτιολογική σκέψη δέλτα υπέρ για το πρώτο τμήμα υπέρ δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται Συγχαρητήρια στον στην κυρία, στην κυρία Τσίμα. Πάμε στην επόμενη έκθεση, Τρτσκόψκι. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, παράγραφος 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια ε, στον κύριο Τρτσκόφσκι. Πάμε στην έκθεση Κάσπαρη, παράγραφος 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται τροπολογία 1 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, Κατά, κατά, ναι. Για το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Το δεύτερο τμήμα απορρίφθηκε. Παράγραφος 8, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίφθηκε. Παράγραφος 11. Υπέρ, κατά, αποχές, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την παράγραφο 11. Έκλεισε η ψηφοφορία και απορρίφθηκε. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Σε ξεχωριστά τμήματα. Ε, η επικεφαλίδα ε, της 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14 σε ξεχωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δε μισό λεπτό. Ε, Μισό λεπτό λέει ο πρόεδρος. Ας προχωρήσουμε. Σας παρακαλώ. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Για το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έκλεισε η ψηφορία. Και εγκρίθηκε. 24. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 34 υπέρ κατά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 34 έκλεισε η ψηφορία απορρίφθηκε 36 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 39. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 43. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για τη 43 ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και εγκρίθηκε. 45. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, αιτιολογική σκέψη Κάπα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη L, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική κλίση, ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση για την πρόταση ψηφίσματος. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίθηκε συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή όρεξη. Κάρο Σούλτς. Πρόεδρε Σούλτς, ε, συγχαρητήρια και καλή όρεξη. Λοιπόν, για την έκθεση ΚΟΠΑ, ο κύριος Μιλάνα έχει ζητήσει το λόγο. Για την έκθεση ΚΟΠΑ.